przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, panie i panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε στις καρέκλες σας, καθίστε στις θέσεις σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego Κυρίσω την επανάληψη της Συνόδου που διεκόπη στις 24 Μαρτίου του 2011. Τα πρακτικά της 23ης και 24ης Μαρτίου έχουν διανεμηθεί και ρωτώ εάν υπάρχουν παρατηρήσεις ως προς τα πρακτικά. Άρα εγκρίνονται. Και θα ήθελα να προβώ σε μια σειρά ανακοινώσεων. Στις 26 Απριλίου θα χαιρετήσουμε, θα θυμηθούμε την 25η επέτειο από το Τσέρνομπιλ. Αποτείουμε λοιπόν, 25 χρόνια μετά, φόρο τιμής στα θύματα αυτής της καταστροφής, σε όσους έχασαν τη ζωή τους, σε όσους αγωνίζονται και ακόμη έχουν ορατά τα σημάδια αυτής της πυρηνικής καταστροφής. Οι αρμόδιες αρχές απέκρυψαν την καταστροφή αυτή από τις, ε, το λαό τους αλλά και από τις άλλες χώρες και εξ αυτού του λόγου κατέστη πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Το Τσέρνομπιλ στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε και αποτέλεσε και υπόδειγμα ε, συνεργασίας μεταξύ κρατών, μεταξύ, μέσα στην διεθνή κοινότητα. Καθώς λοιπόν ε, εορτάζουμε την 25η θλιβερή επέτειο του Τσερνόμπιλ, δεν μπορούμε να μην ε, στρέψουμε τα μάτια και το πνεύμα στο λαό της Ιαπωνίας, της Φουκουσίμα, σε εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ξένους ο σεισμός και το τσουνάμι. Δεύτερη πληροφορία. Πριν από ένα χρόνο στην περιοχή του Σμολένς και στις 10 Απριλίου συγκεκριμένα έχασαν τη ζωή τους μαζί με τον πρόεδρο της Πολωνίας 18 ε, λευτές Πολωνοί και συνολικά 25 άτομα 96 ε, άτομα πολλοί ε, εκ των οποίων ήταν ε, εκπρόσωποι, αξιωματούχοι του κράτους της Πολωνίας. Πολλοί μάλιστα ήταν γνωστοί μου προσωπικοί. Ακόμη δεν είναι γνωστό το υπό ποιες συνθήκες έλαβε χώρα αυτό το ατύχημα, το δυστύχημα. Περιμένουμε να λάβουμε τις τελικές πληροφορίες και αποτείουμε πάλι φόρο τιμής στους οικείους των θυμάτων, στα θύματα και στους οικείους τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εκφράζει την ανησυχία του για την απόρριψη από το Supreme Court των το Δικαστήριων των Πολιτειών της προσφυγής του κυρίου Ντέιβις που ζητούσε αναβολή της εκτέλεσης της θανατικής ποινής Με μία προσφυγή ο κύριος Τρόι Ντέιβις ζητούσε την μετατροπή της θανατικής αυτής ποινής από ε, θανατική σε ισόβια κάθεξη. Αυτό λοιπόν μας θλίβει βαθύτατα. Επίσης ανησυχούμε ιδιαίτερως για τις εξελίξεις στην αρχή του ελεφαντοστού. Οι προεδρικές εκλογές, αντί να εξασφαλίσουν ειρήνη και ευημερία, ε, ε, ρίξαν ε, τη χώρα στο χάος ε, και την αναρχία. Ο Λογόν Μπακμπού δεν ε, δέχθηκε την αναγνώριση της εκλογής του πολιτικού του αντιπάλου και έχει χρησιμοποιήσει κάθε είδου βία για να εξασφαλίσει την επικράτησή του στις εκλογές αυτές. Πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι όποιος είναι υπέτειος για τέτοιου είδους πράξεις βίας θα προσαχθεί στη δικαιοσύνη και σε αυτό θα συμβάλλει μεγάλη του δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν τέλει, όπως σας είχα υποσχεθεί, πρέπει να δώσω ενημέρωση για ζητήματα διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Την Πέμπτη, λοιπόν, και ύστερα από μια συνεδρίαση της Δεσκέψης των Προέδρων, λάβατε μια επιστολή από πλευράς μου σχετική με το ζήτημα αυτό των κατηγοριών περί διαφθοράς εις βάρος ευρωβουλευτών. Λαμβάνουμε λοιπόν αποφασιστικά βήματα για την διατύπωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για τις ομάδες ε, συμφερόντων και τις ομάδες πιέσεως, λόμπι, καθώς και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Προεδρείο το οποίο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα στις 6 για να συστήσει ακριβώς αυτό το θέμα και να λάβει αποφάσεις για, την, για περαιτέρω χειρισμού στην υπόθεση αυτή. Ο κύριος Νίκολσον έχει στήσει το λόγο στην θέση 603. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ στον φόνο την ε, Κυριακή στην Βόρεια Ιρλανδία ενός νεαρού αστυνομικού ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του νωρίς το πρωί. Και δυστυχώς να πω ότι είναι πολλές φορές που έχει χρειαστεί να σηκωθώ εδώ στο κοινοβούλιο. Σε χρόνια είμαι εδώ για να καταδικάσω μια τέτοια πράξη βίας. Νόμιζα ότι έχει περάσει πιο καιρό που θα θρυνούσαμε τέτοια θύματα τρομοκρατίας, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν αληθεύει αυτό. Οι σκέψεις μας λοιπόν συνοδεύουν την οικογένεια αυτού του νέου αστυνομικού που είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Και θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι πρόκειται για μια σαφή ε, και εσκεμμένη πράξη αποσταθεροποίησης της περιοχής μου. Είμαι βέβαιος ότι οι πλειονότητες των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας αρνούνται να επιστρέψουν στο παρόν ή στο μέλλον στα όσα έχουν ζήσει μέχρι τώρα. Έχουν υποφέρει πολλοί οι πολίτες της περιοχής μου και είμαι βέβαιος ότι αυτή η πράξη, ε, αυτός ο φόνος ξυπνά φρικτές μνήμες. Ας απευθύνουμε λοιπόν τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και την ελπίδα ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι έκανα μία δήλωση επ' αυτού του θέματος ε, χθες το πρωί καταδικάζοντας ε, αυτή την πράξη βίας. Ήταν ένας ε, πολύ νέος αστυνομικός και εκφράζω την ελπίδα ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα μπορέσει να ζήσει σε ένα καθεστώς ειρήνης, σε ειρήνη όπως και πρόσφατα. Θα βρείτε την δήλωσή μου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Ντεμπρούν, παρακαλώ. Διαδικαστικό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι δολοφονήθηκε σε μια βομβιστική απόπειρα τρομοκρατική στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Ήταν, πήγαινε στην υπηρεσία του και δολοφονήθηκε ήταν τρομακτικό πλήγμα για εκείνον και την οικογένειά του και όχι μόνο για αυτούς αλλά και για όλα τα άτομα της εκλογικής μου περιφέρειας. Αυτοί που ήθελαν να σταματήσουν την πρόοδο σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, εμείς ε, είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πράξη και θα ήθελα στο Κοινοβούλιο να εκφραστούν τα συλληπιτήριά μας, συλληπιτήρια των μελών του Ευρωκοινοβουλίου στους οικείους του. Και θα ήθελα επίσης να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου εγώ προσωπικά και θα ήθελα να καταδικάσω και καταγγείλω αυτή την τρομοκρατική πράξη. Γκάλαγκερ παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω εσάς γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση καταδίκης αυτής της πράξης εχθές και θέλω να υποστηρίξω τις δηλώσεις Νίκοσον και Ντεμπρόιν εδώ σήμερα Φυσικά εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα, την εγκληματική πράξη, θα πρέπει να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη, η ένοχοι. Η διαδικασία ειρήνευσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέφθηκε με επιτυχία και οι άνθρωποι οι ίδιοι, οι πολίτες της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας καταδίκασαν αυτή τη δολοφονία όσον αφορά τους αστιφύλακες ε, που επλήγησαν και θέλω να επενέσω την θαραλέα δήλωση που έκανε η μητέρα του θύματος ε, για την συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ernst Strasser. Εγκατέλειψε ο Ernst Strasser την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 24η Μαρτίου 2011